εποχές δεκτή. Και περνάμε τώρα σε προφορική τροπολογία της κυρίας Ινφελτ στο εκτιμώντας D. Κυρία Ινφελτ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Ινφελτ. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προτείναμε προφορική τροπολογία να διαγράψουμε αυτή την ε, αιτιολογική σκέψη, γιατί αναφέρεται σε έκθεση που θέλαμε να δημοσιευθεί και δημοσιεύθηκε χθε. Επομένω, είναι περιττή αυτή η διάταξη, κατά τη γνώμη μα. Υπάρχει κανεί που να διαφωνεί με αυτή την προφορική τροπολογία? Αν όχι, ψηφίζουμε τώρα για αυτή την τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, δεκτή η προφορική τροπολογία. Και τώρα ονομαστική ψηφορία για το σύνολο της έκθεσης. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ist geschlossen. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η έκθεση έγινε δεκτή με 581 ψήφους υπέρ. Yeah. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επικονιαστές. Η τροπολογία 2, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 10, ονομαστική ψηφοφορία, Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 12. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και περνάμε αν θέλετε εντάξει, επαλήθευση, παρακαλώ, για την 12. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Παρακαλώ να ε, σηκώνετε καλά το χέρι σας για να βλέπω κι εγώ. Περνάμε λοιπόν τώρα στην παράγραφο 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η παράγραφος 17 του αρχικού κειμένου υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 19, τροπολογίες υπαριθμών 3, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Και περνάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 11, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τέσσερα. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Ως εκ τούτου καταπίπτει το αρχικό κείμενο και περνάμε στην τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Δεκτή. Παράγραφος 27. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Τροπολογία 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η παράγωση 43 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας π σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα Το εκτιμώντας πει πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Περνάμε τώρα στο εκτιμώντας Q, αρχικό κείμενο. Συγγνώμη, τι είπατε. 258 διαδικαστικό. Κοιτάξτε, δεν γίνεται όταν ζητάτε επαλήθευση μετά να το αγνοείτε το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε αυτόν τον τρόπο. Ή όταν κάποιος ζητά επαλήθευση να μην την κάνετε την επαλήθευση. Πρόεδρος, κοιτάξτε, η ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν απόλυτα σαφές. Ως εκ τούτου η ένστασή σας δεν έχει νόημα. Αν εγώ ένιωθα ανασφάλεια, δεν ήμουν σίγουρο για το αποτέλεσμα, θα την επαναλάμβανα την ψηφορία. Πάμε τώρα στο εκτιμώντα Q, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Το 213. Εγώ είμαι στο 113, Πρόεδρε. Από ό,τι φαίνεται ότι δεν είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος συνεδρίασης να αποφασίσει για το ναι ή το όχι γίνεται δεκτή ε, μια τροπολογία. να ζητείται έλεγχος από τους βουλευτές, είναι δικαίωμά εφόσον ε, αναφέρεστε στο κανονισμό και εγώ θα αναφέρω στον κανονισμό και θα σας πω αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου. Πάμε τώρα στο εκτιμώντας ου τροπολογία 1 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτό. Εκτιμώντας AG αρχικό κείμενο υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές Δεκτό. Και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Uh, Προχωράμε τώρα ε, στην διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης. Και ξεκινάμε με την τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 7 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Geschlossen. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 8, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Περνάμε στην παράγραφο 11, Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και περνάμε τώρα στην παράγραφο 12, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές ε, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δε, απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται, τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στην ε, τροπολογία υπαριθμών 4, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Και τώρα έχω μία προφορική τροπολογία του κυρίου Μπράια. Παρακαλώ κύριε Μπράια, έχετε το λόγο. Yes. Thank you. Ευχαριστώ. Βάσει του κανόνα 180 παράγραφος 4 του ιστορικού κανονισμού θα ήθελα να ζητήσω εξ των ε, Πρασίνων μία προφορική τροπολογία στις τροπολογίες 6, 7 και 9 της ομάδας μου για να διορθώσουμε ένα ασφάλμα. Και θα πρέπει αυτές οι τροπολογίες ε, να ανωνυμοποιηθούν. Να διαγραφεί δηλαδή or μην ψευδονιμοποιηθούν, να ανεμοποιηθούν δηλαδή. Προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα ε, ε, του ιατρικού ιστορικού και να αντικατοπτρίζεται και το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά αυτέ αυτές τις ε, τροπολογίες, έχει κάποιος κάτι να πει επ' αυτών. Υπάρχουν αντιρρήσει. Υπάρχει κάποιο που να διαφωνεί. Δεν βλέπω όμω να είναι απαραίτητο αριθμό ανθρώπων βουλευτών που να σηκώνονται, να διαφωνούν. Α, όχι, τώρα βλέπω έχουμε, έχουμε τον απαραίτητο αριθμό όσων διαφωνούν, άρα οι τροπολογίες δεν γίνονται δεκτές. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή την περίπτωση, η βάση του 180 παράγραφος 5 του ιστορικού κανονισμού Εξ ονόματος ομάδας μου θα ήθελα να αποσύρω την τροπολογία, τις τροπολογίες 6, 7 και 9 της ομάδας μου. Ω εκ τούτου, εφόσον 6, 7 και 9 αποσυρθήκαν, πάμε στην ε, ψηφορία 23, τροπολογία 8, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, ε, δεκτή. 24 σε δύο τμήματα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτή για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή παράγραφος 25 αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. να ήταν λίγο οριακό το αποτέλεσμα, γιατί αυτοί που κάνουν το αριστερά δεν σήκωσαν το χέρι τους. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Περνάμε στην παράφορ 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτό. Η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο της έκθεσης υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές δεκτό, το, δεκτή εισήγηση η έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να παρακαλέσω όσους δεν επιθυμούν να προβούν σε αιτιολόγηση ψήφου να βγουν γρήγορα από την αίθουσα για να μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία των αιτιολογήσεων. Σας ευχαριστώ. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου και να ξεκινήσουμε με το ψήφισμα για τις δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων λοαδμό Στον καταλογό μου Έχω την κυρία Μπενιέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ οι ομοφοβικές πράξεις πολλαπλασιάζονται στην κοινωνία μας. Έχουμε προσβολές, επιθέσεις σωματικές ε, και άλλες λόγω του γενετήσου προσανατολισμού φαίνεται σήμερα να θερίζουμε τους καρπούς της πολιτικής σας. Δυστυχώς οι μεταναστευτικές πολιτικές που ακολουθούσατε αποτελούν κίνδυνο ενώ η ομοφιλοφιλία ε, ουσιαστικά ποινικοποιείται με θάνατο σε πολλέ χώρε τη υποσυχάρη Αφρική. Μια γερμανική μελέτη μα έδειξε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ τη ε, ακραίου Ισλαμισμού και τη ε, ομοφοβία. Έτσι ε, λοιπόν ε, μιλάμε για κάποιες περιοχές ε, που ουσιαστικά τίθεται σε περιορισμό λόγω μιας ιδεολογίας. Όμως έχουμε κάποιους ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες αλλά δεν πρέπει να υπερισχύουν αυτά τα δόγματα. Η Κομισιόν τελικά κόβεται το μικρόφωνο. Συγγνώμη, έχουμε αρκετούς ομιλητές. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο σας. Ο κύριος Κέλχερ. Ε, πραγματικά ε, κάποιες πράξεις κρατών ε, μελών κατά των κατοικών ΛΟΑΔΜΟ με έχουν φοβήσει και εγώ υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα όπως μας έχει δείξει η ιστορία είναι τρομερό το να χωρίζουμε μια ομάδα ανθρώπων από κάποιους άλλους όπως και να δημιουργούμε περιοχές χωρίς ΛΟΑΔΜ δηλώνει την άγνοια της ανθρωπότητας οι ΛΟΑΔΜ έχουν το δικαίωμα ε, να χαίρονται τις ελευθερίες, να απολαμβάνουν τις ελευθερίες όπως και η υπόλοιπη κοινωνία. Ε, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους όπως είναι σύμφωνο ε, με το ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ο Ιρλανδικός λαός ψήφισε να καλύπτει ο γάμος και τους γάμους των ομοφιλοφιλών και λοιπόν που στην Ένωση υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται στην ισότητα. Ο κύριος Μπομπάρ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπω ξέρετε φέτο, η Γκαζέτα Πόλσκα, μία από τι ε, κύριε πολωνικέ εφημερίδε που υποστηρίζει την κυβέρνηση, ε, μοιράζει αυτοκόλλητα ζώνε απαλλαγμένε από άτομα ΛΟΑΤΚΙ θέλουν να δηλώσουν ότι έχουν απελευθερωθεί ε, από αυτή την ιδεολογία, όπως λένε. Πρόκειται για μια ε, σταυροφορία κατά της ε, ισότητας όλων των πολιτών, όπως εγκαθιδρύεται στις υπόλοιπες χώρες. Δεν πρέπει η Ευρώπη να αποδεχθεί αυτή την ομοφοβία όταν αυξάνονται οι ομοφοβικές επιθέσεις ακόμα και οι δολοφονίες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καθολικά και αναφέρετα. Όποιος ε, ε, επιτίθεται στα άτομα ΛΟΑΔΜΟΥ, επιτίθεται και στις γυναίκες, στους μετανάστες, στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Η επίθεση κατά ορισμένων δικαιωμάτων είναι πάντα επίθεση και προς τα υπόλοιπα. Φυσικά και υπερψηφίζω αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρίτσι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπάρχουν τα εξή σχόλια από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ της Πολωνίας. Τώρα είναι στη μόδα να είναι κάποιος ε, ενάντια στους ε, ομοφιλόφιλους. Δεν νιώθουμε ασφαλείς. Ε, η νέα εστίαση ε, κατά της ιδεολογίας ΛΟΑΤΚΙ του ε, κυβερνώντος ε, κόμματος στην Πολωνία είχε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα, την ρητορική της κατά των μεταναστών. Μίλησαν κάποιοι για μια φοβία κατά των, της εποσοχάρης Αφρικής. Πάντα έτσι γίνεται με τις φοβίες, ότι κάποιος επιλέγει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό στόχο στον, τον οποίο αντιμάχεται. Έγιναν δηλώσει ε, για τις ε, ζώνες απαλλαγμένε από τα ΛΟΑΤΚΙ και υπόθηκε ότι για μας όλο αυτό με το, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ είναι κάτι το, ε, αφύσικο που προσπαθεί να επιβληθεί στην κοινωνία. Μας είπαν στη συζήτηση ότι οι Πολωνοί ανέχονται την ομοφοβία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κλίμα του μίσου ε, που τροφοδοτεί από τι πολωνικέ αρχέ απέναντι στι κοινότητε ε, ΛΟΑΔ αλλά ε, και προσέγγιση όποιων αιτιολογούν φυσικέ και προφορικέ επιθέσει, είναι απαράδεκτο Εδώ καταστέλλονται τα ευρωπαϊκά δικαιώματα των βελτών και το Κοινοβούλιο, αλλά και η Κομισιόν και το Συμβούλιο πρέπει να τα καταδικάσουν αυτά. Γι' αυτό είμαι υπέρ αυτού του ψηφίσματο, γιατί θα πρέπει τελικά να τεθεί σε εφαρμογή οδηγία κατά τη αγωγή διακρίσεω που εδώ και 11 χρόνια έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο ή να καλύψουμε το νομοθετικό κενό για την προστασία των αδικημάτων βάσει προκατελήψεων ε, λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ε, λόγω φύλου. Τα δικαιώματα των ανθρώπων λάδου είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να τα σέβονται σύμφωνα με τις συνθήκες και τη χάρτα και το διεθνές δίκαιο. Τέτοια ψηφίσματα μας καλούν συνειδητοποιούν ότι ακόμα είμαστε σε κίνδυνο και ότι ακόμη και το δικαίωμα στο νερό πρέπει να το υπερασπίζουμε. Δεν είναι νομοφοβική η Ευρώπη, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. κυρία Σόιντροβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Φυσικά κατανοώ ότι άτομα με αναπηρία έχουν δικαιώματα αλλά και άλλες μειονότητες θα πρέπει να έχουν δικαιώματα που να γίνονται σεβαστά και φυσικά είμαι ακάτε της εισαγωγής διακρίσεως διακρίσεων κατά τον ΛΟΑΔΜ. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό αντίκειται στις βασικές συνταγματικές αρχές και τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι ότι σίγουρα είναι και συνταγματικό στην Πολωνία. Το να διακηρυχθεί ε, μια ζώνη, ζώνη χωρίς ΛΟΑΔΜ, χωρίς ε, την ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ, μπορεί να οδηγήσει σε ομοφοβία και μίσος. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το επιλύσει η Πολωνία. Είναι ερμοδιότητα της Πολωνίας και είμαι σίγουρη ότι οι Πολωνοί πολίτες ε, θα σταθούν κατά της ρητορικής τους μίσους. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δήλωσα αποχή. Ευχαριστώ. Ντάνιλ Χέναν. Ευχαριστώ. Και πάλι έχουμε ένα ψήφισμα που ε, τελικά ε, είναι σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τη μητρότητα και λέμε ότι θέλουμε μια κοινή, μητρότητα, μια κοινή πολιτική για τη μητρότητα. Εγώ πάντοτε θεωρούσα παράδεκτο οι κυβερνήσει να εισάγουν διακρίσεις κατά των πολιτών βάση γενετήσεων προσανατολισμού και στην ε, ε, χώρα μου. Έχω περισπίσει τα δικαιώματα, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτό. Εδώ μιλάμε για την κατάχρηση εξουσίας, για να ευρωπαϊκό γίνει ευρωπαϊκό κάτι, ενώ δεν υπάρχει καμία βάση στις ευρωπαϊκές συνθήκες για εμπλοκή των Βρυξελών. Και ε, τίθεται ξανά και πάλι το ψήφισμα αυτό μόνο ως μία άσκηση, ως ένα εγχείρημα για να ε, πούν ότι αυτοί που δεν το υπερψηφίζουν δεν ενδιαφέρονται για την ομοφοβία. Όχι, δεν ισχύει. Μπορούμε να πιστεύουμε στην ισότητα και αξιοπρέπεια για όλους τους πολίτες, αλλά πρέπει να πιστεύουμε και στη δημοκρατική διαδικασία και στην ηρότητα της κάλπης. Ευχαριστώ, κύριος Τζαμπάσκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εγώ καταψήφισα κατηγορηματικά αυτό το ψήφισμα. Επειδή υποστηρίζει την προπαγάνδα των ΛΟΑΔΜ στην αδερφή μας χώρα, την Πολωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ακόμα χώρες όπου η οικογένεια σημαίνει η ένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός ε, και αποκτούν παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ πιο σοβαρά θέματα να λύσει. Ας επικεντρωθούμε σε εκείνα λοιπόν και ας αφήσουμε τις οικογενειακές αξίες ε, και παραδόσεις ε, στα κράτη-μέλη. Αυτή με το ζόρι επιβολή της ιδεολογίας ε, ΛΟΑΔΜ και της δημογραφικής στρατηγικής μας ε, θυμίζει παλαιότερε εποχέ, όταν οι δικτάτορες έκαναν το ίδιο. Έρχονται τα Χριστούγεννα και τέτοια ιδεολογία είναι απολύτω απαράδεκτη. LGBTIs δεν είναι ιδεολογία των ΛΟΑΔΜ. Έχει να κάνει με τα άτομα. Εγώ ήθελα να μιλήσω για το ψήφισμα και πώς ε, αναφέρεται στην αιμοφοβία, στον αθλητισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, συμβαίνει δυστυχώς. Το ψήφισμα όμως ε, δεν αναφέρει τη σημασία του αθλητισμού στην αντιμετώπιση της αιμοφοβίας. Είχαμε μία πολύ πετυχημένη ε, εκστρατεία στο ποδόσφαιρο εγώ συμμετέχω και στην σχετική ομάδα ε, στον αγγλικό υπόδρομο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις ό,τι αφορά την ε, πολυμορφία και την ισότητα. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Κάποιε φορέ στον αθλητισμό έχουμε πολλέ φορέ φαινόμενα ε, ομοφοβία. Όμω εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στην ισότητα όλων των πολιτών και να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της ομοφοβίας. Η κυρία Φόξ. Εγώ απήχα από αυτή την ψηφορία γιατί λέει ότι θα πρέπει να πενεπικοποιείται ε, το κήρυγμα του μίσους. Αλλά ποιος αποφασίζει τι είναι κήρυγμα μίσους. Παραδείγματο χάνει στο Αρμένο Βασίλειο πάρα πολλοί ε, που αποκαλούνται ε, ομοφοβικοί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται τους ακτιβιστές οι οποίοι απαιτούν ότι εμείς οι γυναίκες πρέπει να αρνηθούμε βιολογικά το σώμα μας, να αρνηθούμε την αυτονομία μας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιβάλλει κάτι σε κράτη στις δημοκρατικές τους αποφάσεις. Ε, ε, δεν τους αρέσει η δική μας ορθόδοξη στάση, δεν τους αρέσουν τα επιχειρήματά μας. Η γραφειοκρατική επιβολή δεν είναι πολιτική νίκη. Το να περάσουν ψηφίσματα δεν σημαίνει ότι κερδίζει κανείς την καρδιά και το μυαλό των ο κύριος Λεμπρετόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισμα, καταψήφισα το ψήφισμα για την Πολωνία γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παρισφρεί στην κοινωνική πολιτική των κρατών μελών. Ε, καταδικάζω και τη διάκριση κατά της Πολωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει στιγματιστεί εξαιτία ε, προγραμμάτων ποινικοποίηση ορισμένων σεξουαλικών ε, τάσεων και εδώ ε, τι καταδικάζουμε, τα αυτοκόλλητα που μοιράζουν κάποιοι δήμοι σχετικά με την ιδεολογία ΛΟΑΔΜΟ. Ε, φυσικά δεν είμαι υπέρ της, ε, των διακρίσεων λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων και προσανατολισμών, όμως θεωρώ ότι εδώ πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Μια κριτική ε, της πολύ λυπηρής αυτής ιδεολογίας του φίλου Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται την Πολωνία και εμείς καταψηφίζουμε ένα τόσο βάναυσο ψήφισμα. Ευχαριστώ, κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Πρόεδρε, εγκρίνοντας αυτό το ψήφισμα κατά της ρητορική μίσους και των δημοσίων διακρίσεων ε, για το κοινωτικό προσανατολισμό, γράφει ιστορία το Κοινοβούλιο και το κάνει όταν πληρούνται δεκαετία από την ε, θέση σε ισχύ τη Συνδίκη Λισαβόνα με τη Χάρτα Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων που απαγορεύει τέτοιε διακρίσει. Θα πρέπει να πω ότι πραγματικά ε, είναι ε, μεγάλο κρίμα να ακούμε στο Κοινοβούλιο ότι πρόκειται για ιδεολογία. Ο γενετήσιο προσανατολισμό δεν είναι η ελευθερία, να ρωτεύεται κανεί, χωρί να υπάρχει διάκριση λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού, αποτελεί μέρο μελλοντών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι λοιπόν η χώρα που δεν το σέβεται, δεν σέβεται το ευρωπαϊκό δίκαιο δίκαιο ε, την στιγμή που έχουμε την επέτειο του Stonewall και χθες μάλιστα ε, γιορτάσαμε χθες ε, την ε, ημέρα ε, για τις αναπηρίες. Πολλά μένουν στην Ευρώπη ε, που πρέπει να απογίνουν. Θα πρέπει να συνεχίζουμε να γκρεμίζουμε διάφορα εμπόδια εισαγωγή σε διάκριση σε διάφορους κλάδους. Όμως αυτό το θέμα που αφορά το γενετήσιο προσανατολισμό είναι ευρωπαϊκό δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τζέκι Τζόντς. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω αυτό το διακομματικό ψήφισμα για τις δημόσιες εκκρίσεις και κατά της λειτουργικής ε, μίσους ε, κατά των ανθρώπων ΛΟΑΔΜΑ και εκφράζω την ελληνική μου στο συνεχιζόμενο αγώνα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίω. Η ενοχή και η συμπερίληψη αποτελούν ε, τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να καταπολεμήσουμε την υπαναχώρηση στα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρος για ζώνες χωρίς δουλειά στην Ευρώπη ή παγκοσμίω. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το ρόλο της εκπαίδευσης στο να προωθήσει υγιείς σχέσεις, στον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίως αυτό ισχύει για τα κορίτσια σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε την ελευθερία της μετακίνησης των ΛΟΑΔΜ, των οικογενειών, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα, ε, όπως έχουν εγγραφεί στο Θεμελιώδη Χάρτη των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων και όχι απλώς θα πρέπει να την προσπίσουμε, αλλά και να τα διευρύνουμε. Πρέπει τους χάρη σε οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών θα πρέπει να έχουμε μελέτη αντικτύπου για το σεβασμό των Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αν αποτυχαίνει να μην υπάρχει συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άντερσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ καταψήφισα αυτό το ψήφισμα γιατί δεν είναι ομοφοβικό. Η παρδοσική οικογένεια από ε, πατέρα, μητέρα και παιδιά είναι νομίζω η καλύτερη και καταψήφισα γιατί για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι εδώ είναι ο χώρο για σοου. Δηλαδή τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων δεν μπορεί κανεί να τα ενισχύσει με το να εκφωνεί πανηγυρικού και να θεσπίζει ψηφίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά με το να ονοματίζονται εκείνοι οι οποίοι καταπατούν τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων και θα του άρεσε πάρα πολύ να του κρεμάσουν ανάποδα. Ε, το θέμα δεν είναι να αρνηθούμε τα δικαιώματα των ομιλοφίλων. Είναι ο πολιτισμός που φέρνουν εδώ στην Ευρώπη και που βιώνουν εδώ τη δολοφονική ομοφοβία. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν όλα αυτά αν πραγματικά παίρνουμε στα σοβαρά υπόψη μας τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Η κυρία Μπρύνα Ανίκα. Ευχαριστώ. Ενώ η καταδίκαση τη βία κατά των ομοφοβικών εξαιτία ε, του προσανατολισμού του θα πρέπει να την χάνει μεγάλη συνένεση ε, και να συμπεριλαμβάνει και ε, τι τοπικέ συλλογικότητε, το σημερινό κείμενο εργαλοποιεί αυτή την επιχειρηματιολογία είναι μια νέα ευκαιρία να επιτεθούμε στην πολωνική κυβέρνηση που δεν πήρε τι φιλελεύθερε αποφάσει που θα θέλατε. Επίσης, καταχρηστικά ε, αναφέρεται το κείμενο στην ομοφοβία ε, κατά της ιδεολογίας ε, ΛΟΑΔΜ. Ε, και κακώς αναφέρει τους λαϊκιστές ως υπεύθυνου ε, ομοφοβικών πράξεων. Ε, και ενώ δεν κάνει καμία σύνδεση μεταξύ της μετανάστευσης και της επιρροής του Ισλάμ και της αύξησης της ομοφοβίας στην Ευρώπη. Ενώ τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια τέτοια σύνδεση. Εμείς καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των ομοφιλοφίλων, όμως δεν θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το θέμα για να προωθείτε τα συμφέροντά σας και να επιτίθεστε στην δημοκρατικά κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Στάνισλαβ Μπρουτζίνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ε, είχα την ε, τιμή ως Υπουργός Εσωτερικών να είμαι μέλος του κόμματος Νομική και δικαιοσύνης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση και αδίκως ε, δέχεται επιθέσεις σήμερα. Άκουσα από την αριστερά ότι η πολωνική κυβέρνηση επιβάλλει διακρίσεις κατά τον ΛΟΑΔΜΟ. Όμως πρέπει να σας πω ότι ω υπουργό Εσωτερικών μαζί με την αστυνομία και άλλες αρχές ε, πάντα προστατεύαμε όσους ένιωθαν απειλή. Ανεξαρτήτως ε, της σεξουαλική ε, ταυτότητα του κάθε πολίτη, όλοι οι πολίτε θα πρέπει να προστατεύονται και οι ομοφυλόφιλοι. Εγώ αισθάνομαι ντροπή ω Πολωνό να ακούω σήμερα όλα αυτά που λέτε. Κάποιοι Πολωνοί από την αριστερά επίσης ακολουθούν τα όσα έχουν υποθεί. Ξέρουν ότι όλα αυτά δεν ισχύουν βέβαια, ότι είναι ψέματα. Κανείς δεν κάνει διακρίσεις κατά τον ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία. Είναι ψέμα. Ευχαριστώ. Αν έχει την καλοσύνη να μην χειροκροτάτε, δεν επιτρέπεται αυτό, δεν προβλέπεται στον κανονισμό. Και περνάμε τώρα στον επόμενο ομιλητή, τον ε, κύριο Μάρτιν Χόργουτ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη στεναρή μου υποστήριξη για το ψήφισμα που πέρασε σήμερα στο Κοινοβούλιο απέναντι ε, στις ΛΟΑΔΜ, ε, στα κηρύγματα μίσους, θέλω να πω στον κύριο Μπριτσίνσκι και σε άλλους, τους φίλους του, ότι ε, πρέπει να επισημαίνονται οι περιπτώσεις στην Πολωνία, όπου ε, βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει επιθέσεις κατά της μεταρρυθμιστικής εκκλησίας της Βαρσοβίας, απλά και μόνο που διώκεται, γιατί έχει προσευχηθεί για την κοινότητα των ΛΟΑΔΜ στην Βαρσοβία. Αυτό είναι ένα είδος δίωξης, το οποίο τελικά δείχνει ότι δεν γίνονται σεβαστές οι αξίες της Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΗ είναι ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να γίνονται σεβαστά. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι προτάσεις ε, ψηφίσματος ε, για δίκαιη φορολογήση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιωμένη οικονομία. Πρώτη έχει το ζητήσει λόγο κυρία Ομπρή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από το 2002 η Apple θα έπρεπε να έχει πληρώσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ προς τους φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λουξ Κέρινγκ της Λοράν θα έπρεπε να έχει πληρώσει 5,2 δισεκατομμύρια παραπάνω. Γιατί αποφεύγουν τη φορολόγηση αυτές τις πολυεθνικές, γιατί θα πρέπει να είναι ηλίθιες για να ε, μην πάνε σε μια χώρα όταν τους ε, εναγκαλίζει. Ε, και η φορολογική παράδοση έχουν καταλήξει σε μια κούρσα προς τα κάτω η Ευρωπαϊκή Ένωση. μάλιστα την ενθάρρυνε. Έχουμε την ε, ιστορική ευθύνη ε, να υπάρχει μεταρρύθμιση των φορολογικών κανόνων στον ΩΣΑ που επιτρέπει στις πολυεθνικές να μην πληρώσουν τους φόρους. Ε, καλούμε να είμαστε φιλόδοξοι με το ψήφισμα αυτό και να υπάρχει ένας ελάχιστος φόρος στις επιχειρήσεις και μια δίκαιη φορολόγηση φορολόγηση ε, στις χώρες όμως ε, χωρίς φορολογική διαφάνεια ή κατάλογο των φορολογικών παραδείσεων οι πολιτικές θα συνεχίσουν να παρακάμπτουν τους φορολογικούς κανόνες και θα πληρώνουν το τίμημα οι πολίτες. Ευχαριστώ κύριο Σπόλτσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός όταν μιλάμε για φόρους και Πολύ σπάνια ψηφίζω για ε, εναρμόνιση στη Φορολογική Ένωση, γιατί εγώ θεωρώ ότι η σημερινή κατάσταση είναι ικανοποιητική. Όμως, δεν θα αρνηθώ την υποστήριξή μας σε αυτό το ψήφισμα. Καταρχήν, γιατί η παραδοσιακή αριστερά έχει προτείνει πράγματα που δεν πέρασαν. Παραδείγματο χάρη τον ε, ελάχιστο ενοποιημένο φόρο. Επίσης, ε, η ψηφιοποίηση της οικονομίας ε, αποτελεί έκκληση δράσης για όλους. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι όλα τα εισοδήματα φεύγουν προς τους φορολογικούς παραδείσους και γι' αυτό καλωσορίζω ε, το ότι την ε, ψηφιακή οικονομία θα πρέπει η Ευρώπη να αντιμετωπίζει στο σύνολό της και γι' αυτό υποστήριξα το ψήφισμα αυτό ενώ δεν το υποστήριξε η αριστερά. Ο κύριος ε, Μίλερ Λέτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστήριξα αυτό το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να καταπολεμήσουμε ε, την δημιουργική λογιστική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη ε, δεν ε, μπορούν να διασφαλίσουν ε, κατάλληλη φορολόγηση της παγκοσμίας ψηφιακής οικονομίας. Όμως θα πρέπει να θέσουμε τέλος στην κατάσταση αυτή όταν οι πολυεθνικές δημιουργούν, γεννούν τεράστια ποσά χρημάτων αλλά δεν πληρώνουν φόρους γιατί έχουν έδρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν υπάρχει ομοφωνία των κρατών μελών στο θέμα αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις διαδικασίες της συνθήκης που να μας επιτρέψουν να ψηφίσουμε σε αυτό με ειδική πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Ευχαριστώ. Ενώ χαιρετίζω την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σε αυτό το νέο κοινοβούλιο για αυτό το σύνθετο ζήτημα, δυστυχώ ε, δεν ήμουν σε θέση να στηρίξω το ψήφισμα. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο λοιπόν το θέμα. Συνεχίζονται διαβουλεύσει σε επίπεδο ΩΣΑ για να βρεθεί λύση για την δίκαιη φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρήσεων. Να ξεκαθαρίσω ότι χαιρετίζω τι προσπάθειε προ ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση. Πρέπει οι εταιρείε να πληρώνουν αυτό που σα αναλογεί. Όμω ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλέ ε, μεγάλε ψηφιακέ επιχειρήσει είναι διεθνεί από τη φύση του. Γι' αυτό συνεχίζω τι ε, ε, συνεχιζόμενες προσπάθειες ε, σε επίπεδο ΣΑ να βρεθεί λύση για αυτό το θέμα μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς. Οι μονομερείς ε, ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προτείνεται σε αυτό το ψήφισμα, θα πλήξει την διεθνή ανταγωνιστικότητα και μπορεί να δημιουργήσει και αντίπεινα από αυτέ τι εταιρείε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένω όμω ανοιχτό και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει επικοδομητικό διάλογο στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα, στο κράτος δικαίου στη Μάλτα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λόπες Αγγιλιάρ. Ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε παρουσία της κυρίας Φορντελάιεν και του κυρίου Σάρλ Μισελ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ενώ γιορτάζουμε τη δέκατη επέτειο της θεσίου ισχύ της Νίκης Λισαβόνας και τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και κάποιοι αναρωτήθηκαν πώ το Συμβούλιο δεν ε, είχε λάβει υπόψη την κατάσταση τη Μαλτέση και άλλοι είπαν ε, γιατί είχε λάβει υπόψη την κατάσταση στην Ουγγαρία ή στην Πολωνία όπου η Κομισιόν πήρε πρωτοβουλία με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο μόνο τρόπο ε, το Συμβούλιο να κάνει τη δουλειά του επειδή το Κοινοβούλιο έκανε τη δική του είναι να υιοθετήσει άπαξ και διαπαντό στο πλαίσιο του Κράτου δικαίου, Δημοκρατία και θεμελιωδών δικαιωμάτων που υιοθετήθηκε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ήρθε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για να έχουμε έναν αντικειμενικό, ρυθμισμένο και τακτικό μηχανισμό ελέγχου και επίσης να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη και να σέβονται το δίκαιο. Το κράτος δικαίου δεν ε, είναι ανεκτό σε μια τέτοια στιγμή που έχουμε περικοπές ε, να ε, λαμβάνουν κονδύλια τα κράτη-μέλη τα οποία δεν σέβονται τους κανόνες περί κράτους δικαίου. Η κυρία Τόμς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. δηλώνω σοκαρισμένη με τις ειδήσει που μας έρχονται από τη Μάλτα σε ό,τι φορά τη διαφθορά και αυτό το φορολογικό παράδεισο. Φαίνεται ότι τα πράγματα και είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φανταζόμασταν. Τα στοιχεία της δολοφονίας της δημοσιογράφου μας οδηγούν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι κάτι το ανήκουστο. Οποιοδήποτε υπεύθυνο πολιτικός θα δηλώνει την παρέτησή του μετά από κάτι τέτοιο. Πριν από δύο χρόνια κάποιοι συνάδελφοι σοσιαλιστέ προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την μαλτέζικη ε, κυβέρνηση και από την άλλη καταδίκαζαν άλλες κυβερνήσεις που δεν ανήκαν στη δική τους πολιτική ομάδα. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν. Ε, διαφθορά, δολοφονίες, ε, αποτυχία του κράτους δικαίου, αυτά συμβαίνουν και αλλού. Επομένως, πρέπει να υπάρχει σωστή τεκμηρίωση οποιασδήποτε διαδικασία κράτου δικαίου με τα ίδια κριτήρια για όλους. Κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Εγώ στήριξα αυτό το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι ο δολοφόνος μιας ε, δημοσιογράφου ε, σε ένα κράτος μέλος, έχοντας κατά νου τις ευρωπαϊκές αξίες, είναι ε, μια απεχθέστατη εγκληματική πράξη και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη Μάλτα, αλλά παρόλα αυτά το κράτος δικαίου και οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν, ως εκ τούτου έχουμε την ηθική υποχρέωση να πούμε ναι, πράγματι ε, θα ελέγχουμε το πώς η πολιτική και η δικαστική εξουσία θα ερευνήσουν την υπόθεση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Μάλτα να εντοπίσουν τους δράστες οι οποίοι θα κληθούν να λογοδοτήσουν στα δικαστήρια και να να τιμωρηθούν ακόμα και αν οι δράστες προέρχονται και από ε, πολιτικούς κύκλους. Μπρουτζίνσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως ε, εγώ στήριξα αυτό το ψήφισμα. Η κατάσταση σε μια δημοκρατική χώρα όπου μια δημοσιογράφος δολοφονείται, μια τέτοια κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να στηρίξει ένα τέτοιο ψήφισμα. Θα αναφερθώ στην παράγραφο 8. Εκεί αναφέρεται ότι αν δεν εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, τότε ισχύει το άρθρο υπαριθμών 7. Έχουμε μια κατάσταση όπου μια δημοσιογράφος δολοφονείται στη Μάλτα ε, και παρεμφερείς καταστάσεις. Έχουμε κάθε μέρα, έχουμε ε, διαδηλώσεις και στη Βαρκελόνη. Η αστυνομία τους εντοπίζει και σε καμία από αυτές τις χώρες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7. Και το άρθρο 7 αφορά μόνο τη δική μου τη χώρα, την Πολωνία, ε, όταν εμείς προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε τη δικαστική εξουσία, η οποία δικαστική εξουσία δεν έχει μεταρρυθμιστεί στην Πολωνία από τότε που είχαμε κομμουνιστικό καθεστώς. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλεχερ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η βιοπικιλότητα. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η επιβίωση της μέλισσας είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, ως νομοθέτες θα πρέπει να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Στη δική μου την χώρα αυτή την εβδομάδα ε, συστήθηκε μία νέα ένωση για να προστατεύσει τη μέλισσα. Η ε, Ένωση των Μελισσοκόμων συστήθηκε για να ε, μπορούν να στηριχθούν οι μελισσοκόμοι, κυρίως εκείνοι που θέλουν να έχουν τις δικές τους τις ε, κυψέλες. Τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι απολύτως απαραίτητο η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική να έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να στηρίζει τους μελισσοκόμους. Και θα ήταν πολύ καλό και εντυπωσιακό αν τουλάχιστον κάθε μέλισσα είχε κάποιον να την προστατεύει. Ευχαριστούμε κυρία Μελά. στήριξα αλλά θέλω να ακούσω τον να του κινδύνω ακόμα πιο πολύ για το πρόβλημα με τους επικοινωνιστές στην Ευρώπη. Υπάρχει πρωτοβουλία της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου του 2018 για τους επικοινωνιστές. Η σημερινή κατάσταση όμως έχει καταλήξει να είναι καταστροφική. Εξαφανίζονται τα σχετικά έντομα κάτι το οποίο απειλεί την ίδια την επιβίωση των κοινωνιών μας, της βιοπικιλότητας γενικά. Η γεωργική παραγωγή εξαρτάται από την επικονίση. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία που μας προσφέρουν οι μέλισσες. Εφόσον εξαφανιστούν, ολόκληρη η οικονομία μας θα καταρρεύσει και πρώτα απ' όλα η γεωργία. Η Κίνα ή άλλες ολόκληρες περιφέρειες θα εξαφανιζόντουσαν χωρίς τις μέλισσες. Επήγε επίσης να ξεπεράσουμε αυτό το κείμενο και να ψάξουμε να βρούμε και την ε, ευθύνη μας, ο καθένας στη δικιά του και να βρούμε λύσεις για την επιβίωση των επικοινωνιαστών. Ευχαριστούμε κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Να επαναλάβω αυτά που είπα και όταν εξετάσαμε την έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή και να υπογραμμίσω ότι με ευρεία στήριξη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε διάφορες προτάσεις για λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εξαφάνισης των μελισσών και των επικονιαστών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε μόνο για τη βιοπικιλότητα, μιλάμε για την ίδια την ουσία, για τους γεωργούς μας, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τη δραστηριότητά τους. Οι επικονιαστές μειώνονται. Και αυτό θα οδηγήσει σε μικρότερη γεωργική παραγωγή. Είναι λοιπόν αναγκαίο να τους στηρίξουμε προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ήπεθρο. Οφείλουμε να προσέξουμε ώστε τα φυτοφάρμακα να αντικατασταθούν από άλλα που δεν καταστρέφουν τις μέλισσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ως ε, σκιώδης ε, εισηγητής ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όλους τους συναδέλφους που υποστήριξαν την πρότασή μας και ενέκριναν αυτό το κείμενο για τους επικονιαστές. Χθε στη συζήτηση ε, ανέπτυξα πολλά επιχειρήματα σε σχέση με το γιατί υπερψήφισα το ψήφισμα αυτό. Εδώ το ζητούμενο είναι να προωθήσουμε το νομοθετικό έργο και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το νέο Green Deal, όχι μόνο στο πλαίσιο της Ευρωβουλής αλλά και ως ιδιώτες. Θα πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, θα πρέπει να αλλάξουμε τις ε, δραστηριότητες μας, τις πρακτικές που έχουμε εφαρμόσει μέχρι στιγμής και αυτό ισχύει και τη σχέση μας και προς τις μέλησες και τους επικονιαστές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βόντρα, ο κύριος Βόντρα Αλεξάνδρου. Ευχαριστώ. Πολύ συχνά λέω ότι πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει να προσέξουμε τα βιαστικά βήματα και τα θεωρητικά ιδεολογικά βήματα. Εδώ και δέκα χρόνια αυτό το κοινοβούλιο ενέκρινε την πράσινη ιδεολογία. Και όσον αφορά την Γεωργία, ο Τσέχος Πρωθυπουργός ε, πλούτησε βάσει αυτού, βάσει του ελαίου κράμβης. Έχουμε παρασιτοκτόνα στα, το ράουντα παραδείγματος χάρη που χρησιμοποιούμε στους κάμπους μας και εκατομμύρια μέλισσες και άλλοι επικονιαστές πεθαίνουν και συνεχίζουν να πεθαίνουν. Γι' αυτό είμαι υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι φταίει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά. Ευχαριστώ και ο και έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι μέλισσες και η ευημερία των μελισσών είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, όχι για μένα και τη χώρα μου τη Βουλγαρία, αλλά και για την Ευρώπη. Γι' αυτό υποστήριξα το σχέδιο ψηφίσματος. Η απαγόρευση των παρασιτοκτόνων είναι πολύ σημαντική αλλά πρέπει να έχουμε και ρεαλιστικές ε, προσδοκίες. Αν δεν βασίσουμε τις δράσεις μας επί της επιστημονικής βάσης, δεν θα είμαστε παραγωγικοί. Υπάρχουν κάποιες ακραίες θέσεις στο κείμενο. Κάποια παρασιτοκτόνα είναι ασφαλή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λογικό τρόπο. Και σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μελέτες, αυτά τα παρασιτοκτόνα δεν είναι επιβλαβή για τους επικονιαστές. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις μέλισσες, μεν, αλλά και τη γεωργία από την άλλη πλευρά, δε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσπης έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα επαναλάβω αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι μέχρι τώρα, ότι εκ πρώτης όψεως το θέμα αυτό φαίνεται να μην ε, ταιριάζει ε, στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό και σοβαρό θέμα, οπότε είναι καλό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με τους επικονιαστές, ασχολείται με την ε, δυνητική καταστροφή από την οποία κινδυνεύει η γεωργία εφόσον χαθούν οι μέλισσες και οι επικονιαστές. Οικονομικά μπορεί να είναι πάρα πολύ σοβαρές οι συνέπειες. Γι' αυτό και στήριξα την έκθεση αυτή, γιατί δεν θέλω να αποδυναμωθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Γεωργία και θα ήθελα να σταματήσει αυτή η καταστροφή. Λε, τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα, τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης. Η κυρία... Μελά. Μελά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας φαίνεται να είναι αναπόφευκτο, διότι η τεχνολογία προχωράει, γνωρίζουμε το σώμα και τη λειτουργία του ακόμα περισσότερο και έχουμε φτάσει μάλιστα σε ένα τέτοιο επίπεδο που η επόμενη επανάσταση δεν μπορεί παρά να είναι ψηφιακή. Κάπου 10% του ΕΠ Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από αυτό τον κλάδο. Το ψήφισμα αυτό λοιπόν, το οποίο στηρίζουμε απόλυτα, αναφέρει τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας με τα δεδομένα ε, για το γεγονός ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα και ότι πρέπει να υπάρχουν και ρήτρες εξασφάλισης.